την 3η Ιουλίου επαναλαμβάνεται. Τα πρακτικά τη συνεδρίασης τη 3 η Ιουλίου διατίθενται. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ενστάσεις. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά.